προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δύο μάλλον προφορικές ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Γκάλαγκερ. Πέντε λεπτά, ο οποίος όμως δεν είναι εδώ, οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Καντέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Επίτροπε, θέλησα να υπάρξει η συζήτηση για την προστασία του λαβρακιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί συζητάμε για την επιβίωση του είδους αυτό. Είναι ένα ευγενές αλίευμα υψηλής οικονομικής απόδοσης το οποίο ε, ζητούν και αυτοί οι οποίοι αλλιεύουν ερασιτεχνικά και οι επαγγελματίες. Στην μάχη και στον Ατλαντικό ε, είναι σημαντική η μερίδα της αλληλείας από τους ε, επαγγελματίες les pêcheurs récréatifs pratiquant eux la traque de surface γρηγροί παραγάδια και ε, Οριμάζει ε ε, ε, ε, αναπαραγωγικά τον τρίτο ή τον τέταρτο χρόνο της ζωής του και φτάνει τα 30 με 40 εκατοστά. Η αναπαραγωγή γίνεται μετά από μία μακρά περίοδο συνάντησης των αλλιευμάτων με μεγάλη πυκνότητα ε, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εκεί φυσικά τα αλλιεύματα είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Ε, η προστασία των ειδών ανήκει στις χώρες ε, μεμονωμένα και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γαλλία πήρε κάποια μέτρα στα πλαίσια της Επιτροπής για την Προστασία των λαβρακιών. Σαν παράδειγμα μείωση της αλλιευτικής δραστηριότητας στην αναπαραγωγική εποχή 100 μέτρα τουλάχιστον ε, για ε, τα παραγάδια και περιορισμός ποσοτικός ε, σε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Πρόκειται για τολμηρά μέτρα αλλά ανεπαρκή. Για την ερασιτεχνική αλληλεία αποφάσισαν να αυξήσουν εθελοντικά το μέγεθος, το ελάχιστο της αλίευσης, αποδεικνύοντας ότι συνειδητοποιούν την ανάγκη προστασίας του είδους αυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα αυτό και να το οργανώσει σε κοινοτικό επίπεδο. Τα προγράμματα του 12 μας δείχνουν ότι υπάρχουν προβλήματα για το μέλλον του είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχε προταθεί μείωση 20% ανάμεσα στο 2008 και το 2012. Η γνωμοδότηση της ΙΦΡΕΜΕΡ του 2011 δημιουργεί αμφιβολίες για την επιβίωση του είδους και αυτή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στα κράτη-μέλη να παρακολουθήσουν τις συνέπειες των δραστηριοτήτων των αλλιευτικών επαγγελματικών και ερασιτεχνικών έτσι ώστε να επιτραπεί η αηφορία στην εκμετάλλευση του είδους. Αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην απαγόρευση αλίευσης του λαβρακιού, αλλά στη σωστή οργάνωση. Μέτρα διαχείρισης που θα επιτρέψουν στους αλίες να ασκήσουν τις δραστηριότητές τους στα πλαίσια των ποσοστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις και στα πλαίσια μιας πολυετούς ε, μορφής διαχείρισης ελέγχοντας τα αλλιεύματα, την ποσότητά τους, ελέγχοντας επίσης και ε, την εμπορία του είδους που έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Ε, δεν θα πρέπει επίσης ε, να περάσουμε σε λεπτομέρειες ή μάλλον θα πρέπει να περάσουμε σε λεπτομέρειες για περιορισμούς της ερασιτεχνικής αλληλείας ορίζοντας το ελάχιστο μέγεθος και το, μεγάλο, το μέγιστο ε, ποσό, εν πάση περιπτώσει, ε, ε, ηχθείων που μπορεί να αλλιεύουν. Και θα πρέπει να περιμένουμε επίσης και την έκθεση του 14. Θα ζητήσω από την Επιτροπή να δημιουργήσει και τάκ ποσοστώσεις στην αλίευσή του σε αιτήσια βάση και θα πρέπει να αυξηθεί στα 40 εκατοστά το ελάχιστο ε, μέγεθος μήκους του ψαριού που να επιτρέπεται προσαλίευση. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά για την προστασία του λαβρακιού. Έτσι μόνο οι αλληλείς θα συνεχίσουν να εκμεταλλεύονται αυτό το υψηλής προστιθέμενης αξίας αλίευμα και θα συνεχίσουν και ε, οι δυνατότητες που παρέχει η αλληλεία αναψυχής. Λοιπόν, πολιετές πρόγραμμα στην Μάχη και τη Βαλτική. Ευχαριστούμε κύριε Καρντέκ. Το λόγο έχει τώρα ο δεύτερος συντάκτης προφορικής ερώτησης, ο κύριος Γκάλαχερ. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ισλανδία και οι Φερόες ε, αλλιεύουν σκουμπρί αδιακρίτως τα τελευταία χρόνια. Η Ισλανδία μάλιστα μονομερός α, αύξησε τα αλλιεύματα από 1% το 2006 στο 23% την αλλίευση σκουμπριού το 2013 σε είδατα μάλιστα που το απόθεμα αντιμετωπίζει δυσκολίε και οι Φερόες από 4,6% το 2009 αύξησαν σε 23% την αλλίευση σκουμπριού το 2013 και πάλι στην ίδια περιοχή όπου έχουμε προβληματικά αποθέματα. Χθε το απόγευμα στο Λονδίνο, μετά από επανειλημμένες συναντήσεις, βρέθηκε τελικά συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Νορβηγίας και νησιών Φερόων σε ό,τι αφορά την αλίευση σκουμπριού στον βορειοανατολικό Ατλαντικό. Μάλιστα είχαμε ε, εδώ και πολλά χρόνια περιμένω αυτή τη συμφωνία. Βέβαια η Ισλανδία αποχώρησε από τις συνομιλίες, δεν έχει προσυπογράψει τη συμφωνία και έχει καθορίσει μονομερώς ποσοστώσεις για το 2014. Το μέγιστο επιτρεπόμενο αλίευμα που προβλέπει ε, η χθεσινή συνεδρίαση είναι 1,2 εκατομμύρια τόνοι για το επόμενο έτος που ανταποκρίνεται στην ε, σύσταση της ΆΙΣΙΣ για αύξηση του γενικού ΤΑΚ. Είναι για μας θετική αυτή η εξέλιξη. Ε, οι, οι ποσοστώσεις μας από 57.000 τόνους θα πάνε στους 105.000 ε, τόνους ε, για τομέα μάλιστα που έχει τζίρο 155 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα έχουμε σημαντική αύξηση, δηλαδή 6% αύξηση στις, προ, στις προσωρινές ποσοστώσεις που είχαμε ακούσει στις αρχές του έτους. Βέβαια, μακροχρόνια Ανησυχούμε για το 12,6% ποσοστό στη, στην αλίευση που έχουν λάβει τα νησιά Φερόες, που είναι αδικαιολόγητο ποσοστό υψηλό και θα οδηγήσει σε απώλειες του ευρωπαϊκού ελευτικού κλάδου και κυρίως του ιρλανδικού ελευτικού κλάδου. Πάντως, χαιρετίζω την ε, πρωτοβουλία της Επιτρόπου Δαμανάκη που θα πρέπει να αναλάβει την πλήρη ε, κατάσταση και τη, ήταν πολύ ισορροπημένη διαχείριση που έκανε του όλου θέματος ε, αλλά δυστυχώς ήταν απογοητευτική η απογοητευτικό το αποτέλεσμα και μάλιστα η απουσία της κυρίας Δαμανάκη σήμερα δείχνει πόσο σέβεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Επίτροπος και κυρίως την Επιτροπή Αλίας γιατί φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν έτοιμη να καταλήξει συμφωνία πάση θυσία με οποιοδήποτε αίτημα και ε, ήταν έτοιμη να δεχτεί να πάει από το 9 μέχρι το 12%. Δεν είχε ε, δυστυχώς τα μέσα να επιβάλλει κυρώσει στις χώρες αυτές όταν η συντριπτική πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τάχθηκε υπέρ της επιβόλης κυρώσεων. Δυστυχώς δεν το έκανε αυτό η Επιτροπή. Πάντως ευτυχώς υπήρχε στις διαπραγματεύσεις η Νορβηγία που ε, επέμεινε και ουσιαστικά βοήθησε τον ευρωπαϊκό κλάδο. Χρειαζόμαστε μακροπρόθεσμη λύση για τη βιωσιμότητα των αλληλευμάτων σκουμπριού και των αποθεμάτων σκουμπριού, ε, σημαντικός τομέας και για την αλληλεία και για τη μεταποιητική βιομηχανία. Βέβαια, το νέο καθήκον ε, για τη συνέχιση της κατάστασης θα ε, ανατεθεί στον νέο επιτρόπο. Ελπίζουμε να τα καταφέρει καλύτερα. Ούτως ή άλλως και το προσφυγάκι Νορβηγίας ε, έτυχε υπεραλίευσης και γι' αυτό κατέρευσε το σχετικό απόθεμα. Ε, ελπίζω να μην έχουμε αντίστοιχη περίπτωση και με τα αποθέματα σκουμπρίου, γιατί η περίπτωση του, με το ψάρι προσφυγάκι της Νορβηγίας και την ε, κατάρρευση αυτού του αλλιεύματος μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί μπορεί να συμβεί και σε άλλα αλλιευτικά αποθέματα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων οι κυρώσεις κάτι που ούτως ή άλλως υπερψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πριν τις ε, θερινές διακοπές, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε μας ε, κοίταξε κατάματα και μας υποσχέθηκε ότι θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα και θα επιβάλλει και κυρώσεις. Και τι έκανε, τίποτα απολύτως δεν έκανε η Επίτροπος. Και μάλιστα φαίνεται ότι υιοθέτησε μια πολιτική πισόπλατη για την Νορβηγία και εις βάρος των συμφερόντων του ευρωπαϊκού κλάδου. Ευτυχώς όμως η Νορβηγία στάθηκε αμετάκλητη στις διαπραγματεύσεις, γιατί η Ισλανδία δεν είναι συνεργάσιμη από όπως είπατε τις διαπραγματεύσεις. Και το Μάιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε ε, το μέτρο αυτό κατά των νησιών Φερόες ε, για την αλήψη ε, βατραχόψερου και άλλων ψαριών, θα πρέπει τώρα να επιβληθούν κυρώσει και στην Ισλανδία και μάλιστα με άμεσο αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λεβαντόσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ξεκινήσω από την διατήρηση των αλλιευμάτων του Λαβρακιού. Εμείς συζητάμε το θέμα λοιπόν αυτό με σας από το 2012. Από τότε είχαμε δύο εξελίξεις. Από τη μία έχουμε τώρα πλέον περισσότερες επιστημονικές, επιστημονικά ευρήματα σχετικά με την δυνατότητα ειφορίας. Και δεύτερον έχουμε τη μεταρρύθμιση της ε, κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Τα επιστημονικά σταχεία ε, δείχνουν μειωμένη βιομάζα και απαιτούν να αλλιεύονται λιγότερα λαβράκια γενικότερα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται τις επιστημονικές αυτές παρατηρήσεις και τις υποστηρίζει. Σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής έχουμε περάσει στη φάση τώρα της περιφερικοποίησης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει πλέον να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αναπτύξουν τους εθνικούς τους έλεγχους σε ένα πρόγραμμα ολοκληρωμένο για την προστασία του είδους. Πρόκειται για μια διαδικασία εκ των κάτω προς τα άνω η οποία λαμβάνει υπόψη νομίζω όπως και εγώ τις παρεμβάσεις που προηγήθηκαν. Πάντως η λογική της μεταρρύθμισης της κοινή αλλιευτικής πολιτικής είναι η περιφερικοποίηση. Πρέπει λοιπόν να την πραγματοποιήσουμε και να την ελέγξουμε αν λειτουργεί. Αυτό θα μας επιτρέψει να ελέγξουμε την ποιότητα των ε, εθνικών στοιχείων και θα ζητήσουμε από την επιστημονική κοινότητα εάν τα εθνικά μέτρα είναι επαρκή ή όχι θα υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη, αλλά επαναλαμβάνω η λογική της μεταρρύθμισης της κοινή ε, αλλιευτικής πολιτικής είναι η περιφερικοποίηση. Όπως ζήτησε και ο κύριος Κάντεκ, υπάρχει πάντα η δυνατότητα, υπάρχει η επιλογή να λειτουργήσουμε και σε κοινωνικό επίπεδο, σε κοινοτικό επίπεδο αλλά πολλά κράτη-μέλη είναι εναντίον αυτής της λογικής και είναι υπέρ της περιφερικοποίησης σε εθνικό επίπεδο κάτω ακριβώς από τις διαχειριστικές δυνατότητες των ιδίων των κρατών μελών. Έτσι έχουν λοιπόν τα πράγματα. Από τη μία έχουμε τη λογική των επιστημονικών στοιχείων, από την άλλη την περιφερικοποίηση και λαμβάνω επίσης υπόψη και την παρέμβαση του κυρίου Καντέκ, ο οποίος ζητά να υπάρξει και μια διαφορετική λογική για ευρωπαϊκές ποσοστώσεις. Προς το παρόν όμως δεν τίθεται το θέμα αυτό γιατί η πλειοψηφία των κρατών μελών είναι εναντίον αυτής της λογικής. Για το σκόμβρο τώρα. Και εδώ συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πάνω από τέσσερα χρόνια για να βρούμε μια κάποια λύση. Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν μετακινήσεις και αλλαγές σε στάλιεύματα και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ευαισθησίες ορισμένων θυγωμένων κρατών μελών. Έχουμε κάποια στοιχεία και το μήνυμα το οποίο θα έπρεπε να είναι θετικό, χθες καταφέραμε να συμφωνήσουμε, όπως είπε και ο κύριος Πατ Γκάλαγκερ, ε, υπήρξε συμφωνία με την Νορβηγία και τις νήσους Φαρόες, χωρίς όμως την Ισλανδία. Η Ισλανδία τελικά έμεινε εκτός της συμφωνίας. Αυτό ακολούθησε πολλές εξαντλητικές διαπραγματεύσεις με τις υπόλοιπες χώρες και δεν συμφωνώ με αυτούς που είπαν ότι δεν λάβαμε υπόψη μας εμείς τα βέλτιστα των συμφερόντων των αλλιέων των κοινοτικών και την αηφορία των αλλιευμάτων που είναι και αυτό η άλλη πλευρά του νομίσματος. Έχουμε τώρα μία συμφωνία μπροστά μας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Έχουμε ένα προβλέψιμο μέλλον για τον έλεγχο των αλλιευμάτων του σκόμβρου στον Ατλαντικό. Τώρα και εξ ονόματος της συναδέλφου κυρίας Δαμανάκη η μη συμμετοχή της Ισλανδίας είναι απογοητευτική. Μία από τις επιλογές είναι οι πιθανές κυρώσεις, αλλά νομίζω ότι σήμερα θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να προωθήσουμε ε, το ε, καλό μήνυμα του ότι έχουμε κάποιες προοπτικές αηφορίας, αηφόρου εκμετάλλευσης με δύο χώρες που εμπλέκονται στην Αλία και αυτό είναι καλά νέα στους Αλίες της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπολείπων κοινοτικών χωρών. Η πρωτοβουλία πάντα είναι στην πλευρά μας, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα λάβω σοβαρά υπόψη αυτά τα οποία θα μου πείτε και αυτά τα οποία θα πούν και τα υπόλοιπα μέλη ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βασικό είναι ότι σημειώνεται η συμφωνία με τις δύο χώρες, ε, με την Ισλανδία όχι και ε, ακούγονται φωνές για επιβολή κυρώσεων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάτο Τροβέρ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια και πρόκειται για κοινή συζήτηση, θα επικεντρωθώ στο σκουμπρί, γιατί ο κύριος Καντέκ ε, μίλησε για το λαβράκι. Λυπούμε για την απουσία της αρμόδιας Επιτρόπου Αλία. Μάλλον εκείνη θα πρέπει να λυπάτε, γιατί είναι από τις λίγες φορές που έστω και μερικώς θα μπορούσα να της δώσω συγχαρητήρια για την χθεσινή συμφωνία με τις παράκτες χώρες του Βορειοανατολικού Ατλαντικού. Η χθεσινή συμφωνία με ε, αναγκάζει να αλλάξω κάπως την ε, χθεσινή μου την ε, ομιλία που είχα ετοιμάσει χθε και μάλιστα με ιδιαίτερη χαρά. Όπως αναφέρθηκε το πρόβλημα της αλίας κουμπουριού δεν είναι καινούριο. Είχαμε πολλές πρωτοβουλίες και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδειξε η όβια υπομονή για το θέμα αυτό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν έγραφα την ομιλία μου ε, προβληματιζόμουν από, με διάφορα θέματα. Γιατί, λέω, μετά από ένα τρίμηνο δεν έχουμε καταλήξει συμφωνία για τα οριστικά τάκτα, μέγιστα επιτρεπόμενα λιεύματα. Ιδιαίτερα για το σκουμπρί, η καθυστέρηση αυτή θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Επίσης, διαρωτήθηκα, γιατί η Ισλανδία και τα νησιά Φερόες μονομερός ε, ε ενέκριναν κάποια τάκ και ποσοστώσεις για το σκουμπρί ε, αδιαφορώντας για τους υπόλοιπους εταίρους και κυρίως για την Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε πολύ συγκαταβατικοί απέναντι σε ορισμένες χώρες ε, που δεν συμμορφώνονται, ενώ σε άλλες είμαστε πολύ αυστηροί. Γιατί λοιπόν έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Η επίτευξη συμφωνία ε, είχε θεμελιώδη σημασία, αλλά όχι πάση θυσία, όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Είναι πολύ μερική η συμφωνία ε, έχουμε μια αύξηση του, της ποσόστοσης. Εμείς πρωτοστατήσαμε στην Ισπανία και επίσης πρωτοστατήσαμε κατά της παράνομης αλίας και της επιβολής κυρώσεων. Υπάρχουν όμως προβλήματα. Το θέμα της Ισλανδίας και της αποχώρησης από τις διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δείξει πυγμή και αποφασιστικότητα και καμία συγκαταβατικότητα απέναντι ε, σε χώρες που δεν συμμορφώνονται. Έστω και αν αυτή η χώρα είναι η Ισλανδία. Ευχαριστώ. Κύριε Μάτο Αντροβέρ, ε, θέλει κάποιος να σας υποβάλει ερώτηση με γαλάζια κάρτα. Τη δέχεστε, ο κύριος Ρούμπιχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ομιλητή, διότι βεβαίως για μας η Ελία έχει πολλές επιπτώσεις στην Ευρώπη και με ενδιαφέρει να μας πει ποια είναι τα πλονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της συμφωνίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες ψαράδες και κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις που μεταποιούν τα ψάρια. Θεωρείτε ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε έχει πλονεκτήματα και μήπως έχει και κάποιο μειονέκτημα. Νομίζω ότι την ερώτηση σας θα πρέπει να την απευθύνετε στην Επίτροπο. Κατά τη γνώμη μου είναι ικανοποιητική η συμφωνία. Τώρα για τις επιμέρους χώρες, για την Ισπανία είναι θετική. Έχουμε αύξηση για το, της ποσότητες πάνω από 40.000 τόνους. Οπότε οι αλλιές θα έχουν κάποια βεβαιότητα για το τι δικαιούνται να αλλιεύσουν. Τώρα, για τις μεμονωμένες χώρες τους εκτιμήσεις είναι διαφορετικές. Αλλά σίγουρα η ερώτηση αυτή καλύτερα να αποταθεί στην Επιτροπή και όχι σε μένα. Είναι σε θέση να απαντήσει καλύτερα από μένα. Κύριε Ρόντουστ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Μερικές φορές ε, τα γεγονότα και η επικαιρότητα τρέχουν πολύ πιο γρήγορα από την ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου. Χαίρομαι λοιπόν πάρα πολύ που επιτεύχθηκε συμφωνία για τη διαχείριση του σκουμπρίου και χαίρομαι πάρα πολύ ε, κυρίως ε, για τους αλλοί στη Βόρεια Ευρώπη οι οποίοι επλήγησαν από τη σύγκρουση που εμένετο. Παρά λοιπόν αυτά τα ευχάριστα πρέπει να ασκήσω και κριτική το γεγονός ότι ο πόλεμος για το σκουμπρί διήρκησε τέσσερα χρόνια, αυτό είναι δυσάρεστο για όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Και δεν είναι καλό παράδειγμα αυτό για τη διεθνή ελεία, δεν είναι καλό το ότι οι γείτονες και συνεργάτες στη Βόρεια Ευρώπη δεν μπορούν να συνεργαστούν. Από τέτοιου είδους συγκρούσεις κανείς δεν ε, κερδίζει και τελικά ε, παραμένουν ε, ζημιωμένοι μόνο οι ψαράδες, αλλά βεβαίως και το περιβάλλον. Η σύγκρουση με την Ισλανδία και τη νήσους Φερόε επεκτάθηκε ακόμα και στην Βαλτική, οι ε, ψαράδες της Ρέγκας ε, επλήγησαν γιατί δεν μπορούσαν να αποκτήσουν πιστοποιητικά. Όσο δεν υπάρχει βεβαίως ε, συμφωνία ανάμεσα στη Νορβηγία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αποθέματα. Η Νορβηγία ε, ήθελε τη συμφωνία αλλά μόνο με την Ισλανδία. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δεν τολμώ να πω ποιο ήταν σκληρό ή ποιο έπρεπε να ενδώσει πρώτο. Όμω, τολμώ να πω ότι χρειαζόμαστε κατεπηγόντως διεθνείς οργανισμού έτσι ώστε τέτοιου είδου θέματα να τα επιλύουμε με δίκαιο τρόπο και ξεκάθαρα. Το σκουμπρί δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τελευταίο ψάρι που αλλάζει βιότοπο ε, και γι' αυτό ε, θα πρέπει να βρούμε μια λύση. Σε αυτή τη θητεία πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες οι οποίες ε, θα οδηγήσουν την βελτίωση της ε, διαχείρισης των αποθεμάτων. Πρέπει να είμαστε περισσότερο παρόντες και πρέπει επίσης να ε, συνεργαζόμαστε με βουλευτές από την Νορβηγία και την Ισλανδία και το ίδιο ισχύει και για τους συνεργάτες μας στο Νότο. Εμείς οι βουλευτές εκπροσωπούμε το λαό και οι πολίτες δεν θέλουν το πόλεμο του σκουμπριού αλλά θέλουν μια λογική πολιτική. Για ένα λεπτό κυρία Μπαραντίκα. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να, ήταν εδώ η κυρία Δαμανάκη να τη, για να τη συγχαρούμε, γιατί θα ήταν δίκαιο να το κάνουμε για τη συμφωνία ε, στην οποία κατέληξε με την Ορβηγία και τις Φερόες. Αλλά θέλουμε περισσότερη συμμετοχή, περισσότερη διαφάνεια και επιστημονική τεκμηρίωση για να, για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την Ισλανδία. Είναι απαράδεκτο μονομερός η Ισλανδία να αυξάνει τις ποσοστώσεις της. Από το 2000... Ε, έχει αυξήσει κατά 23% το, την αλίευσή της. Δεν ανεχόμαστε ε, ο, ο ελευτικός στόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα βασικός, να μην έχει αρκετές ποσοστός για να μπορεί με βιώσιμο και αποδοτικό τρόπο να συνεχίσει την αλίευση. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα κάνετε απέναντι στην Ισλανδία, θα επιβάλλετε τελικά κυρώσεις ή όχι. Και θα ήθελα στα πλαίσια του ε, ελέγχου που ασκείτε να ρωτήσετε την Ισπανική κυβέρνηση με την νέα ποσόστοση που έχει για τους 40.000 ε, ε, τόνους ε, σκοπεύει να κατανείμει το ποσοστό που χρειάζεται ο βασικός στόλος που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αλία σκουμπρίου. Ευχαριστώ κύριε Λέβιν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι και ευχαριστώ και Επίτροπε. Οι κλιματολογικές αλλαγές είναι μια πραγματικότητα και ξέρετε ότι ο σκόμβρος ε, είναι ένα παράδειγμα ε, σύγκρουσης για αλλιεύματα και φυσικούς πόρους γενικότερα ε, που θα συναντήσουμε στο μέλλον. Έχουμε και άλλα προβλήματα, έχουμε μετανάστευση ειδών, έχουμε πλημμύρες, έχουμε αλλοιώσει στο κλίμα και απαιτείται αλληλεγγύη και μηχανισμοί για σωστή εκμετάλλευση των πόρων που είναι διαθέσιμοι. Πώς μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στον τομέα του σκόμβρου γενικότερα μετά από τις μετακινήσεις των κοπαδιών προς το βορρά. Οι λύσεις που δώσαμε δεν ήταν πολύ καλές. Το 2013 μας είχαν πει ότι η κατάσταση των δεδομένων και των στοιχείων που είχαμε στη διάθεσή μας ήταν εξαιρετικά κακή. Δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα ουσιαστικά. Μόνο δύο στόλοι μας είχαν δώσει στοιχεία για τις απορρίψεις και ακριβώς λόγω της έλλειψης αυτών των στοιχείων υπήρχε μια συστηματική ε, παρανόηση της κατάστασης και δεν υπήρξε γενικά καμία ουσιαστική πρόταση και για την αηφορία ε, της εκμετάλλευσης των αλλιευμάτων. Πρέπει να βρεθεί μια δίκαιη λύση λοιπόν με τις Φερόες, ε, την Νορβηγία και την Ισλανδία. Θα πρέπει ταυτόχρονα όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους για το τόσο σημαντικό αυτό αλίευμα που βρίσκεται σε κακή κατάσταση και μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο άμεσα. Η έλλειψη αδιφορία στην εκμετάλλευση των αλλιευμάτων είναι απαράδεκτη και θα πρέπει να αυτοπεριορίσουμε τις ανάγκες μας και θα πρέπει επίσης στους στόλους οι οποίοι δεν παρέχουν στοιχεία σχετικά με τα παλιεύματα και τις απορρίψεις να μην έχουν πρόσβαση στην αλλιεύση του συγκεκριμένου είδους. Ευχαριστώ. Στίβενσον ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρε, καταρχήν πιστεύω ότι είναι άδικο να επιτίθεται κανείς την κυρία Νταμανάκη για το ότι δεν βρίσκεται εδώ. Είπε στη διάσκεψη των Προέδρων ότι έπρεπε να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη σε αυτή τη συνδιάσκεψη για τα διεθνή αποθέματα. Ε, βεβαίως, ε, θα μπορούσε να υπάρχει κάποια ευελιξία να τις επιτρέψουν να βρίσκεται εδώ για αυτή τη συζήτηση. Ξέρω πως και ο κύριος ε, Γκάλαχαρ δεν επιτύχαμε καμιά μεγάλη ρήξη 12,6 της ποσόστοσης ε, το δώσαμε στις νήσους ε, ε, Φερόες και 16,5% τα προβλέπουμε για την Ισλανδία και τη Ρωσία ελπίζοντας ότι αργότερα θα προσχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία. Νομίζω είμαστε πάρα πολύ γενναιόδοροι. Και ο λόγος που το κάναμε είναι γιατί οι ICS μας λένε ότι μειώθηκε κατά πολύ ο γόνος και έχουμε τώρα 1,2 εκατομμύρια τάκ το οποίο ήταν διπλάσιο από από ό,τι πριν από δύο χρόνια. Αυτό ίσω όμω να μην είναι αηφόρο και εντωμεταξύ ενδέχεται να ζημιωθούμε. Αυτό είναι νομίζω μια ευχάριστη είδηση και θα χαροποιήσει όλους. Ο κύριος Φεραίρα παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όπως ε, αναφέρει το ψήφισμα που θα ψηφίσουμε εντός ολίγου, οι κλιματικές, περιβαλλοντικές και άλλες συνθήκες επηρεάζουν τον τρόπο μετανάστευσης των αλληλευτικών ειδών καθώς και την κατανομή των πληθυσμών των ψαριών. Η κατανομή λοιπόν των ποσοστώσεων θα πρέπει να παρακολουθεί αυτές τις αλλαγές στη σχετική αυθονία των ε, αλληλευτικών ειδών. Και επίση θα πρέπει να στηρίζεται σε ενημερωμένη επιστημονική ε, τεκμηρίωση για την κατάσταση του αποθέματο και το, τη σχετική κατανομή του πληθυσμού. Και αυτό θα πρέπει να ισχύει και για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ε, τρίτες χώρες, αλλά και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τα ληφτικά είδη του βορειοανατολικού Ατλαντικού, θα πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την κατανομή των ποσοστώσεων μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντα υπόψη τα επιστημονικά στοιχεία. Η εξέλιξη του αποθέματο οδήγησε, για παράδειγμα, στην Πορτογαλία σε μεγαλύτερη σχετική αυθονία του σκουμπριού στα εθνικά χωρικά ύδατα τα τελευταία χρόνια. Η ποσόστοση όμως που ισχύει δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Αυτό αποδεικνύει και το γεγονός, το γεγονός ότι ε, ε, εμείς ε, αξιοποιούμε πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο νωρίς ε, την ποσόστοση εξαιτίας της αυθονίας ακριβώς του αλληλευτικού πόρου. Θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν απόψε αυτά τα στοιχεία και οι αλλαγές στα αποθέματα και στην παρουσία του πληθυσμού των ψαριών. γιατί αυτή η σχετική σταθερότητα θα πρέπει να οδηγήσει σε μια απόλυτη σταθερότητα που θα, δεν θα ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και θα είναι άδικη. Ο κύριος Κιούν για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Επίτροπε Λεβαντόφσκι, Αν πάμε πίσω στο 2009 θα, θα πούμε όλοι ότι τότε η Ισλανδία ήταν ε, στο χείλος ε, της επτόχευσης και ε, αγωνιζόταν. Εμείς είπαμε λοιπόν με σαφείς ε, προϋποθέσεις ε, τι ε, μπορούμε να προσφέρουμε αυτά τα ιδιαίτερα δικαιώματα τα οποία είχε επιτρέψει στον εαυτό τη. Ε, θα έπρεπε από αυτό να γίνουν διαπραγματεύσεις το 2010 οι Ισλανδοί ε, παραβίασαν όλες τις συνθήκες αλίευσαν 130.000 τόνους σκουμπρίου και έτσι λοιπόν το σκουμπρί πλέον κινδυνεύει στην περιοχή το ότι και τώρα και πάλι δεν παρίστανται αυτό δείχνει ότι ακολουθούν το δικό τους δρόμο και εμείς ε, πρέπει να τους επιπλήξουμε. Δεν πρέπει να υποφέρουν όλοι οι άλλοι στόλοι. Το ότι τώρα υπήρξε μια συμφωνία με τις νήσους Φερόε και με την Νορβηγία, αυτό είναι ιδιαίτερα θετικό, παρότι βέβαια πρέπει να δούμε και τους συγκεκριμένους αριθμούς, να δούμε ε, ποια θα είναι τα αποθέματα ε, και οι ποσοστώσεις μάλλον που χορηγούνται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως αυτό που έχει σημασία είναι ότι καλό που επιτύχαμε συμφωνία με την Νορβηγία. Η Νορβηγία επίσης είναι πάρα πολύ καλό το ότι γνωρίζει πολύ καλά τι θα συμβεί με το σκουμπρί, με τις ε, ποσοστώσεις της ε, και μετά να δούμε λιγάκι τι θα γίνει με τη Βαλτική θάλασσα, Σκάγκερα, Κακάκεγκρατ ε, ή να δούμε και τι θα γίνει με τη Ρέγκα Τώρα λοιπόν εφόσον συμφώνησαν οι Νορβηγοί έχει ανοίξει ο δρόμος ε, και ε, θα μπορούν να αλλιεύουν με βάση την αρχή MSY της μέγιστης απόδυσης. Ε, στο μέλλον ισχύει και η άλλη αρχή MSC, η πιστοποίηση. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πιστοποιούμε τα ψάρια μας και να έχει και καλύτερο μέλλον το δικό μας το κρατήδιο, το Mecklenburg-Vorpommern. Το αποτέλεσμα τέλος πάντων που επιτεύχθηκε νομίζω ότι είναι θετικό Ευχαριστώ κύριος Σάντζες Πρεσέδο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Το 2015 ίσως θα είναι η χρονιά που θα σταματήσει ο πόλεμος του Σκουμπριού. Γιατί η ελλείψη αυτού του είδους εδώ και χρόνια ήταν ε, ε, επίμαχο και τα τελευταία χρόνια εκατοντάδες ε, αλείς της Γαλλικίας για γρηγρή έκαναν διαδηλώσεις εξαιτία ε, των χαμηλών ποσοστών που έχει η Ισπανία και το Σκουμπρί. Με τη συμφωνία ε, επιτέλους ε, αποκαθίσταται μια βεβαιότητα και μια προβλεψιμότητα και μια πιο ακριβωδική κατανομή των ποσοστώσεων. Μια σωστή κατανομή μεταξύ των παρασυρώμενων πλαδιών και των γρηγρή. Επίσης, με την Ορβηγία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περίπου το 90% ε, των αλληλευμάτων. Ε, Είναι απαράδεκτο λοιπόν για το 2013 η Ισλανδία και οι Φερόες να μονοπολούν σχεδόν το 50%. Ε, χαιρόμαστε για την συμφωνία που ε, χθε στο Λονδίνο και να αφήσουμε ανοιχτή την πόρτα της διαπραγμάτευσης για να την προσυπογράψει αυτή τη συμφωνία και η Ισλανδία. Ε, χάρη στην Ορβηγία αυξήθηκαν κατά 60% τα αποθέματα το 2014, κατά 64% συγκεκριμένα, και χάρη σε αυτό θα μπορούσαμε να έχουμε και διμερή συμφωνία με την Ορβηγία για το σύνολο του αλληλευτικού κλάδου. Τώρα θα πρέπει τα κράτη-μέρη να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Ό,τι αφορά το λαβράκι, ε, θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάγνωση κατάστασης ολευτικού αποθέματος για να υιοθετήσουμε τα κατάλληλα μέτρα. Σας ευχαριστώ κυρία Κάρη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την συμφωνία που, που στην οποία κατέληξε χθε. Ήταν πολύ σημαντική αυτή η συμφωνία η κοινή αλληλευτική πολιτική πολλές φορές είναι ε, παράλογη από άποψη και οικονομική και βιωσιμότητας ε, των αλληλευτικών αποθεμάτων. Γιατί μερικές φορές όταν ζητούμε αύξηση της αλλήλευσης ε, με το επιχείρημα της αύξησης των αποθεμάτων δείχνουμε μια υπερβολική απληστία. Παρακαλώ Ευχαριστώ κύριε Φανίστελ Ροϊ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαίρομαι λοιπόν για τη συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, ιδιαίτερα στο όνομα των αλλιέων που ενδιαφέρονται άμεσα. Πρόκειται για μια καλή προοπτική η οποία ανοίγεται ε, για όλους. Η συμφωνία με την Ορβηγία προβλέπει ακριβώς να υπάρξει μια σταθεροποίηση της κατάστασης. Τώρα, σχετικά με το λαβράκι, υπάρχει μια προφορική ερώτηση η οποία έχει προβλεφθεί. Είναι σαφές ότι απαιτούνται μεγάλες αλλαγές στην παρούσα φάση. Όταν μας λέει ο Επίτροπος ότι υπάρχει μια αποκεντρωμένη περιφερικοποιημένη πολιτική που θα λύσει το πρόβλημα, αυτό δεν είναι απάντηση είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ε, διαχείριση μακροπρόθεσμη του προβλήματος και η πρωτοβουλία του κυρίου Καντέκ ακριβώς αυτό κάνει έτσι ώστε να υπάρξει τελικά στο τέλος μια αηφόρος αλία η οποία να μπορέσει να διατηρήσει το αλίευμα για πάρα πολλά χρόνια. Απαιτούνται λοιπόν αλλαγές και ακριβώς ε, λόγω αυτών που είπε και ο κύριος Καντέκ πρέπει να έχουμε περισσότερες επιστημονικές πληροφορίες και στοιχεία. Ο κύριος Καντέκ μας μίλησε για τη συμφωνία αυτή. που απαιτεί τεχνικά στοιχεία και επιστημονικά στοιχεία αποτελεσματικά, πλούσια, που θα επιτρέψει να γίνεται σωστά ο έλεγχος. Η επικουρικότητα καλή είναι, αλλά πού είναι τα αποτελέσματα. Πρέπει λοιπόν να διευκρινίσουμε προς την αρμόδια επίτροπο, την κυρία Δαμανάκη, ότι έχουμε κάποια καλά νέα στον τομέα του σκόμβρου, αλλά τα αποτελέσματα για το λαβράκι θα πρέπει να επανεξεταστούν. Ευχαριστώ. Τόμας, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συνάδελφοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ε, μια ιστορική κίνηση στη διαχείριση των αλλιευτικών πόρων ε, με την μέγιστη αηφόρο ε, δυνατότητα αλλιεύσης. Αυτό θα πρέπει να συνοδευτεί από διαχειριστικά μέτρα καλύπτοντας τις ανάγκες και των εταίρων μας. Τίθεται το θέμα της αλλιείας αναψυχής. Από το 6 μέχρι το 10 η επαγγελματική αλληλεία έφτανε τους 5.000 τόνους και η αναψυχή 2.300 τόνους. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι μορφές διαχείρισης δεν είναι ικανοποιητικές. Θα κάνει λοιπόν μια νομοθετική πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριλαμβάνοντας και την ερασιτεχνική αλληλεία. Νομίζω ότι τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής δεν μπορεί να αγνοηθούν και δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο στους επαγγελματίες αλληλείς. Θα πρέπει επίσης να επιβάλλουμε τα μέτρα που παίρνουμε εμείς και στους εταίρους μας. Ο αγώνας για περισσότερα αλλιεύματα της Ισλανδίας και ε, των υπολείπων χωρών θα θίξει φυσικά ε, τα αλλιεύματα. Τώρα για τα είδη τα οποία δεν υφίστανται ε, ποσοστώσεις η τελευταία αριθμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα λιεύματα στην Μεσόγειο δείχνει ότι δεν υπάρχει τελικά συσχετισμός ανάμεσα στην αλλιευτική δραστηριότητα και την επιβίωση του ίδιους. Νομίζουμε ότι η έννοια της αηφορίας πρέπει να εφαρμοστεί σε όλους. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Θα, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Φράγα. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή για τη χθεσινή συμφωνία του Λονδίνου. Και μάλιστα με τη συμφωνία αυτή ευνοούνται οι Ευρωπαίοι αλείς και ε, είναι ένας κόλαφος για αυτούς που ασκούν παράνομη όπως είναι η Ισλανδία. Ελπίζω στο μέλλον να προσυπογράψει τους ε, κανόνες για μια βιώσιμη και νόμιμη ελεία. Οι δεμοί υπάρχουν νομικοί μηχανισμοί και μπορούμε να τους ε, εφαρμόσουμε για να επιβάλλουμε κυρώσει. Απευθύνω λοιπόν έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το λάβει υπόψη. Πάντω χαίρομαι για τη χθεσινή συμφωνία. Οι Ευρωπαίοι αλληλεί που βρισκόταν σε οριακή κατάσταση εξαιτία ε, τη πάνη του αποθέματο ε, σκουμπριού, με τι ποσοστώσει αυτέ ε, θα αναπνεύσουν επιτέλους οι αλληλείς. 136% αύξηση είχαμε στην ποσόστοση σε σχέση με το 2013 ε, και έτσι ε, θα γίνει η κατανομή μεταξύ των διαφόρων ειδών αλίας, όπως είναι το γρηγρί, παραγάδια, μηχανότρατες και ούτω καθεξής. Έτσι επιλύονται τα πολύ σοβαρά προβλήματα που μας ταλάνιζαν μέχρι τώρα για το σκουμπρί. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επιτροπέ. Σήμερα το πρωί χαιρετήσαμε τη συμφωνία που επιτέχθηκε χθε στο Λονδίνο μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση τη Νορβηγία και των Ίσων Φερό. Γιατί υπήρχε ε, ανεύθυνη αλία και έπρεπε να τελειώσει καλή συμφωνία, υπάρχουν όμως ε, προβλήματα και όσον αφορά τα πλεονεκτήματα η Ισλανδία δεν θα πάρει μεγαλύτερη πρόσβαση στα δικά μας τα ύδατα. Αυτό είναι καθοριστική σημασία για να προστατευτεί η αγορά για τους Ιρλανδούς ε, ψαράδες και για τους Ιρλανδούς πάλι ε, καλά τα νέα πάνω από 60% η αύξηση σε 150.000 τόνους γιατί το σκουμπρί για την Ιρλανδία είναι ένα πολύτιμο ψάρι. Όπως και οι άλλοι και εμείς ανησυχούμε όσον αφορά την αύξηση του στόκ ε, της ε, ποσόστασης που δίνεται στις νήσους ε, Φερόες. Αυτό μας ανισχύει πραγματικά. Πάντως είναι θετικό το ότι επιτεύχθηκε η συμφωνία γιατί αυτή θα επιτρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις για ανεύθυνους ψαράδες και για αυτούς που δεν τηρούν τη συμφωνία. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που θέσατε τα θέματα. Εγώ ήρθα εδώ να υπερασπιστώ φυσικά τη χθεσινή συμφωνία. Είναι μια ισορροπημένη συμφωνία που δημιουργεί ένα σταθερό πλαίσιο για την αλία. Και φυσικά για την Ισλανδία οι εξελίξεις είναι απογοητευτικές. Ε, ίσως θα πρέπει να γίνει μια επιπλέον προσπάθεια πριν περάσουμε στη συζήτηση των κυρώσεων. Τώρα, ε, το θέμα των μονομερών δράσεων της Γρυλανδίας ε, είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί, που δεν αναζητεί ακριβώς ε, την ιδιότητα της παράκτιας χώρας. Η κυρία Δαμανάκη είναι σε μια πολύ σημαντική συνάντηση και ζητά συγγνώμη αλλά είπε ότι ε, στην επόμενη ευκαιρία, στη συνάντηση με την Επιτροπή Αλίας θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Ε, τώρα για το λαβράκι, τα αποτελέσματα από ό,τι καταλαβαίνω δεν είναι απόλυτα δεκτά. Ε, η λογική της περιφερικοποίησης δηλαδή και των εθνικών ευθυνών για τη διαχείριση των ελέγχων αλίευσης. Ακούω κάποιες φωνές εδώ, όπως άκουσα και για τις κυρώσεις για την Ισλανδία για τα μη συμβατικά εμπλεκόμενα μέρη για το σκουμπρί, όπως επίσης και για ευρωπαϊκές ποσοστώσεις σαν επιλογή πλέον για το λαβράκι. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κλείνει η συζήτησή μας για τα θέματα αλίες. Πριν περάσω στο επόμενο θέμα πρέπει να σας κάνω κάποιες ανακοινώσεις. Οι αρμόδιες γερμανικές αρχές ε, ε, μου ε, ανακοίνωσαν τον ορισμό της κυρίας Ανέτ Κόβιους αντικαταστώντας τον κύριο Λένε. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφο